Okay. Welcome to Καλώς στην Επιτροπή όλοι σας. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω όλους του εκπροσώπους των Εθνικών κοινοβουλίων σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με ε, του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής εφαρμογή των προτεραιοτήτων με την έκθεση πρωτοβουλία που έχουμε για τις προτεραιότητε του 2012. Αυτή ε, η συζήτηση εντάσσεται συνεδρία συντακτική της Επιτροπής μας. Δεν είναι ούτε διακοινοβουλευτική, ούτε κοινή με άλλη Επιτροπή. Αλλά καταβάλλονται προσπάθειες να ενισχυθεί η συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι ε, πραγματικά επίκαιρο να κάνουμε μια συζήτηση για, το 2012 γιατί ε, οι ε, συστάσεις αναχώρα που ενέκρινε το Συμβούλιο πριν τις νέες διακοπές καλούνται ε, να εφαρμοστούν στα σχέδια των προπολογισμών που συζητούν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επιπλέον, ναι, μαζί με την κρίση και την κρίση χρέους που επηρεάζει την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, η απόφαση που θα ληφθεί από το εκάστοτε κοινοβούλιο ε, για τον προπολογισμό του 2013 μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη. Μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας λοιπόν για τον κύκλο του 2012 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον εισηγητή, τον κύριο Ζαμπόλ Γκοζές. Στόχος της συζήτησης αυτής είναι μεταξύ άλλων να τροφοδοτηθεί από τη συζήτηση πριν εγκριθεί η έκθεση αυτή τον Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, αναφέρουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κύκλο 2012 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πριν με τη σειρά τη εκείνη η θέση της οικονομικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία για το 2013. Διαδικαστικά, 22 γλώσσες έχουμε. Ελπίζω ο καθένας να βρει τη γλώσσα του για τους εθνικούς βουλευτές σήμερα έχουμε κάρτες αν θέλετε να ζητάτε το λόγο για να διευκολυθεί η συζήτηση. Παρακαλώ. Συμπληρώστε μια κάρτα που θα ζητάτε το λόγο και δώστε τη σε ένα κλητήρα. Ε, οι ευρωβουλευτές θα σηκώνουν το χέρι τους ως συνήθως για να σας αναγνωρίζω. Και επειδή σας γνωρίζω, θα δώσω πρώτα το λόγο στον Ζαν να κάνει την παρουσίαση της έκθεσης του. Μια δέκα λεπτά περίπου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεσή μου αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Να υπενθυμίσω ότι η δημιουργία του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συνδέθηκε με την διαπίστωση ότι οι χώρες της ζώνης ευρώ βιώνουν μία περίοδο στα πλαίσια της οποίας οι μορφές συντονισμού της οικονομικής πολιτικής τους είναι ανεπαρκής και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλές κρίσεις, ιδιαίτερα την κρίση του δημοσίου χρέους. Η ιδέα είναι μέσω του εξαμήνου να περιορίσουμε τις μεταδοτικές κινήσεις από τη μία χώρα στην άλλη λόγω των αντιφάσεων των δημοσιονομικών και των οικονομικών πολιτικών των χωρών αυτών. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέψει σε επίπεδο ευρωπαϊκό να γίνει μια συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες της πολιτικής τους, της δημοσιονομικής και της οικονομικής και στο εσωτερικό τους, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, έτσι ώστε και αν αυτό ε, χρειαστεί να υπάρξουν οι απαιτούμενες διορθώσεις το εξάμεινο αυτό, το οποίο <clears throat> διαρκεί άνω των έξι μηνών βέβαια, αλλά έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη να χρησιμοποιούμε λέξεις που δεν λένε τίποτα στον πολίτη. Το εξάμεινο αυτό είναι το πρώτο τμήμα λοιπόν του προπαρασκευαστικού έτους του προϋπολογισμού, με μια ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών για να εξετάσουν τις συνθήκες στα πλαίσια των οποίων προετοιμάζονται τα σχέδια εθνικών προϋπολογισμών. Και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε σωστά τα στοιχεία τα οποία σε συγκεκριμένους προϋπολογισμούς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αρνητικά στις γειτονικές χώρες και τις λεγόμενες μεταδοτικές αυτές συνέπειες. Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λοιπόν γίνεται και ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στην προπαρασκευαστική φάση εκφέροντας την γνωμοδότησή του για τις συστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προταθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παρεμβαίνει στην κατάσταση της κάθε χώρας. Αντίθετα προσπαθεί έτσι ώστε η μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται να λειτουργεί αποτελεσματικά και ε, ιδιαίτερα σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο να είναι επακριβείς, σαφείς και αποτελεσματικές. Δεν χρειάζεται να επαναλάβει κανείς γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις του είδους απαιτούνται ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Για να είναι αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να περιλαμβάνει συστάσεις οι οποίες να στοχεύουν τις καταστάσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα και για τις οποίες καταστάσεις απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις. Το δεύτερο έτος του χρόνου είναι το λεγόμενο εθνικό εξάμεινο θα μπορούσαμε να πούμε. Εκεί τα κράτη-μέλη συνεχίζουν όπως ακριβώς έχουν συνηθίσει θα έλεγα για τη διαμόρφωση των δημοσιονομικών τους καρτών στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους, της προετοιμασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις οι οποίες έχουν γίνει δεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ βέβαια τίθεται το θέμα του αμοιβαίου βάρους, θα έλεγα, των μεν και των δε. Δηλαδή, ε, τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κοινοβουλίων των κρατών μελών και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό. Η έκθεση με την οποία με επιφορτήσατε λοιπόν είναι σε φάση προπαρασκευαστική. Κατετέθη ένα κείμενο πρώτο προετοιμασίας Ακούσαμε τις απόψεις των συναδέλφων, εργαστήκαμε πάνω στο κείμενο ήδη και προχθές, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες των ΜΕΝ και των ΔΕ, έτσι ώστε οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του εξαμήνου να είναι θέσεις και ρεαλιστικές και να αποδεικνύουν την πραγματική επιθυμία του Κοινοβουλίου στο δικό του επίπεδο να εμπλακεί στην διαδικασία αυτού εξαμήνου. Στο δικό του επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή δημοκρατικού ελέγχου προς το Συμβούλιο. Θα πρέπει εδώ να, να αποσύρουμε από μπροστά μας την δυνατότητα μιας παρανόησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει να αυτό ανακηρυχθεί ως κριτής των συστάσεων που απευθύνονται προς τα κράτη-μέλη, ούτε και να αντικαταστήσει τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων. Απλά επιθυμούμε σε επίπεδο αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρώπη να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος να ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο σχέδιο εκθέσεως λοιπόν το οποίο υποβάλλω προς συζήτηση και προς εμπλουτισμό από τους μεν και τους δε εγώ έχω κρατήσει την αντίληψη που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικά με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και σχετικά με την αναζήτηση της βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα των εθνικών προϋπολογισμών. Το θέμα είναι βέβαια εάν τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σεβασθούν τα στοιχεία της πολιτικής τα οποία θεωρούν και ανακοινώνουν προς τα έξω ότι θα βελτιώσουν την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει και είναι επίσης σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των μέτρων αυτών και να προχωρήσουμε στην επαναξιολόγησή τους με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί. Θεωρούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό το να προτείνει κανείς συνεχώς νέα μέτρα, χωρίς τα μέτρα τα οποία εκ των προτέρων έχουν αποφασιστεί δεν έχουν πραγματικά τεθεί σε λειτουργία και αξιολογηθεί σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Αυτά λοιπόν ήταν πάρα πολύ σύντομα τα στοιχεία που δείχνουν πόσο διαφθρώνονται η έκθεση αυτή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για τις ε, υπηρεσίες των κρατών μελών. Να πως πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρηματοπιστωτική διατήρηση για να καταλήξουμε σε μια σταθερότητα απαραίτητη για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω τώρα πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση. Ε, είναι ένα ε, το λόγο ένα λάξ. Δύο ευρωβουλευτές πρώτα. Μάλλον όχι, δύο βουλευτές Εθνικό Κοινοβουλίο και μετά ένας ευρωβουλευτής. Γιατί περισσότεροι εθνικοί βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Τρία λεπτά είναι ο χρόνο αγόρευση και παρακαλώ να τον τηρήσετε, γιατί έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Αν θέλει να μιλήσει πάνω από ένα βουλευτής από μια χώρα, παρακαλώ συντονιστείτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια μεταξύ σα. Γιατί σε τελική ανάλυση Ε, αν θέλετε, επειδή θα μιλήσουν δύο εθνικοί βουλευτές, το δεύτερο γύρο να μιλήσει ο δεύτερος από την ίδια χώρα στην αρχή, να ακούσουμε από διαφορετικές χώρες. Και μετά ο εισηγητή θα συνοψίσει σύντομα. Από Εθνικά Κοινοβούλια, λοιπόν. Ο κύριος Καϊαν Κρένε, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών από την Αυστρία και από τη Σουηδία στη συνέχεια ο κ. Καλ Χάμιλτον. Ο κ. Δεν ξέρω πού είστε παρακαλώ. Three minutes. Thank you, Madam Chair. Um, and thank you for... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά, ο κύριος Κράινερ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση ε, της έκθεσης του. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω στα γερμανικά γιατί μου είναι πιο εύκολο. Το πρώτο θέμα ευρωπαϊκό εξάμεινο έναντι εθνικού εξαμήνου. Τα κοινοβούλια εργάζονται όλο το χρόνο και για το προϋπολογισμό και δεν μπορεί να αναχθεί αυτό σε ένα εξάμεινο μόνο και μας στην Αυστρία οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται την Άνοιξη ε, γιατί έχουμε τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα και καθορίζονται οι βασικές γραμμές για την επόμενη τετραετία κάθε φορά από την Άνοιξη. Γι' αυτό ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εγώ το βλέπω ως ένα έργο ε, και εργαλείο παρακολούθησης όχι βραχυπρόθεσμο αλλά μέσο και μαχροπρόθεσμο για να μπορεί κανείς να συγκρίνει πώς ε, αναπτύσσονται τα κράτη-μέλη σε σύγκριση το ένα με τον άλλο. Βεβαίως σε διαδικασίες μεταρρυθμίσεων καταλαβαίνω ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ε, ούτε από το ένα έτος στο άλλο φαίνονται μέσω στα αποτελέσματα. Είναι μέσω μακροπρόθεσμες οι εξελίξεις εκεί και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε τέτοιες προσδοκίες ότι μετά από ένα εξάμεινο αμέσως μπορεί κάποιος να κάνει ε, την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή των συστάσεων 100%. Ούτε είναι ο στόχος αυτός. Ε, βασικό είναι να επικεντρωθούμε στο στόχο, όχι στο δρόμο. Γιατί μέχρι τώρα... Ε, Είχαμε επικεντρωθεί στο στόχο, ενώ τελευταία αρχίζουμε και κολλάμε στο δρόμο, στον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Νομίζω θα πρέπει να παραμένει αυτό στην εθνική αρμοδιότητα, ο δρόμος που θα οδηγήσει στο στόχο αυτό. Να συμφωνούμε τους στόχους ευρωπαϊκά, αλλά ε, κάθε χώρα να επιλέγει το δρόμο που θα την οδηγήσει εκεί. Γιατί μέχρι τώρα έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία από τη μια και τα χρηματοπιστωτικά και από την άλλη ε, τα κοινωνικά και τα εργασιακά. Και τώρα και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο κάνει σκέψεις να μετατοπίσει αυτή την ισορροπία. Όχι. Εγώ το θεωρώ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα κοινωνικά και τα οικονομικά. Και ένα τελευταίο, το πιο σημαντικό, βλέπουμε τους στόχους το 2020 και τα λοιπά, 40-50 σημαντικούς στόχους προσπαθούν τα κράτη-μέλη να τους πληρώσουν, αλλά αυτή τη στιγμή το 3% ε, το έλλειμμα και το 60% του χρέους κυριαρχούν. Και στη συζήτηση είναι μεγαλύτερες προτεραιότητες από κάποιες άλλες. Βεβαίω είναι σημαντική στόχη και καλό είναι που προσλαμβάνουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος, αλλά, αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ε, παραμερίζεται, που είναι η ενεργεία και κυρίως η ενεργεία των νέων, που είναι περίπου ε, εξίσου σημαντικό στόχος και είναι και πάρα πολύ εύγλωτος για τη λειτουργία μιας κοινωνίας. Και όταν συζητούμε για υπερβολικά ελλείμματα, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε υπερβολική ανεργία και ιδιαίτερα υπερβολική ανεργία των νέων, το τονίζω. Και πιστεύω ότι εδώ πραγματικά ε, δεν είναι μόνο η πολιτική συζήτηση αλλά και η ουσιαστική ε, λειτουργία θα πρέπει να προσανατολίζεται και στην ανεργία των νέων. Όχι, δεν υποτιμώ καθόλου το έλλειμμα και τα λοιπά, αλλά εξίσου σημαντικό είναι η ανεργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάμελτον, τρία λεπτά. Microphone. Yeah. Εγώ προέρχομαι από την ε, Σουηδία που δεν ανήκει στο ευρώ. Ορισμένοι από εμά θέλουμε να μπει στο ευρώ η Σουηδία κάποτε, άλλοι όχι. Αλλά και για τα δύο πλευρές αυτές βουλευτών είναι σημαντικό να είναι ανοιχτέ οι πόρτες ώστε να μπορούμε αργότερα να μπούμε στο ευρώ ή σε κάποια άλλη ρύθμιση σε σχέση με την οικονομική πολιτική. Έχουμε πολύ αυστηρό σύστημα εποπτείας του προϋπολογισμού. Όχι επειδή είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι, απλά επειδή μας τύπησε μια κρίση πολύ σοβαρή τραπεζική χρήση στις αρχές της δεκαετίας του 90, πολύ πριν από τους υπόλοιπους ε, εθνικοποιήσαμε τις τράπεζες, αλλά αργότερα πουλήθηκαν εκ νέου σε ιδιώτες. Τώρα έχουμε λοιπόν ε, ειδικό κανονισμό για τον προϋπολογισμό που εισήχθη τότε πολύ αυστηρό 1% στόχο πλεονάσματος όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, πολύ συγκεκριμένους ε, οικονομικούς δείκτες και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πώς θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Έχουμε επίσης στόχους ονομαστικούς όρους ε, όσον αφορά τα μελλοντικά όρια δαπανών και αυτά καθώς και άλλα μέτρα όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού συστήματος τότε μας ε, ωφέλησαν πάρα πολύ έκτοτε. Είμαστε λοιπόν υπέρ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και όλων αυτών των δικτών και στόχων που θεσπίζονται μέσω αυτού καθώς και υπέρ της εξέτασης των χωρών και των σχολείων και συστάσεων. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν θέλουμε άλλες χώρες ή κομισιόν να έχει άποψη όσον αφορά το μισθολόγιο τον, στην ε, Σουηδία είναι αποκεντρωμένο και λειτουργεί καλά το σύστημά μας στη Σουηδία. Ε, γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών και δεν θέλουμε καμία ανάμειξη εκεί. Επίση, αυτό το φθινόπωρο θα ληφθεί η απόφαση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και θα συζητήσουμε στην Επιτροπή φυσικά την Τραπεζική Ένωση καθώς και το τμήμα της εποπτείας που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το πακέτο. Εν γέννη λοιπόν το πρόβλημά μας είναι όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι η ανεργία των νέων και η ανεργία που έχει φτάσει στο 7,3 ή 4% αυτή τη στιγμή. Και δουλεύουμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό και όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά όπως είπα θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαστε υπέρ αυστηρών ε, κανόνων δημοσιονομικής εποπτείας. Σας ευχαριστώ. Η Ελίζα τώρα. Θα ακούσουμε πρώτα τους σκεώδεις εισηγητές. Η Ελίζα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ελίζα Φερέιρα, σας ευχαριστώ. Εγώ Είμαι σκιώδης εξ ονόματος των Σοσιαλιστών Δημοκρατών για την ε, έκθεση που αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ευχαριστώ για τη συνεργασία και το ανοιχτό πνεύμα του συναδέλφου κυρίου Μποζές. Ήθελα να υπογραμμίσω εδώ το εξή. Αυτή η πρόταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα καθορίσει την ισορροπία και θα αφήσει την ελευθερία στα κράτη-μέλη να ορίσουν το μέλλον τους μέσω του προπολογισμού τους και από την άλλη πλευρά θέτει κάποια όρια στην ελευθερία αυτή που επιβάλλονται από το ότι έχουμε κοινό μέλλον ε, διασύνδεση αλεξάρτηση των οικονομιών μας, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μία από τις απαντήσεις στην κρίση, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως η κρίση προέκυψε μετά από 12 χρόνια, κυρίως ε, ε, στην Ευρωζώνη, ανεπάρκειας και διαρκούς και αυξανόμενης ανισορροπίας ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών μελών. Και αυτό το στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη εφόσον θέλουμε να διορθώσουμε τις εκδηλώσεις της ίδιας αυτής της κρίσης που σχετίζονται με το χρέος και το έλλειμμα. Η ανάπτυξη και η απορρίθμιση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών επέφερε στην πραγματική οικονομία αντίκτυπο που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι χώρες. Στόχος είναι λοιπόν αυτή η εναρμόνιση αυτή τη στιγμή και αυτό ε, η διαδικασία η δημοσιονομική να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την πειθαρχία που επιβάλλεται από το πακέτο των 6 μέτρων και από το πακέτο των 2 μέτρων αλλά και μέσω της μεταρρύθμισης του πόνου λοιπόν για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη, αλλά και μέσω μια σύνθεση ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη σύγκληση ανάμεσα στι οικονομίε των κρατών μελών, όλο ιδιαίτερο αυτών τη Ευρωζώνη, και επιπλέον μια σύνθεση ισορροπημένη ανάμεσα στου στόχου ε, για καινοτομία, επιστήμε, έρευνα, ε, τεχνολογία μέσα στην ατζέντα 2020, αλλά και αύξηση της απασχόλησης μέσα, στα, μέσα από τα ίδια μέτρα. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν εργαζόμαστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αναγνωρίζοντα ότι στι συστάσει τη η ίδια η Κομισιόν θα πρέπει να επαληθεύσει σε ποιο βαθμό ε, επιτυγχάνονται οι στόχοι που είχαν προβληθεί και να είναι έτοιμη να διορθώσει τι ίδιε τι συστάσει όταν αυτέ δεν λειτουργούν ή δεν δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή τα προβλεπόμενα αποτελέσματα γιατί είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ο ρόλος των κοινωνικών φορέων σε κάθε μια από τις χώρες μας, των συνδικάτων, της ε, κοινωνικής διαβούλευσης, πέρα από την επαφή με τους εθνικούς ε, βουλευτές και τους τοπικούς ε, ερετούς άρχοντες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα εργαζόμαστε ώστε να βρούμε κοινή βάση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Από τη Γαλλική Γερουσία, ο κύριος Μαρινή, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων. Από το Βέλγιο, ο κύριος... Συγγνώμη, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά, λέει πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα θα μιλήσει ο κύριος με Μαρινή από τη Γαλλική Γερουσία. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Μαρινή έχει αρχίσει την ομιλία του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση μετά από τη συνάντηση που είχαμε τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Στις απαντήσεις που είχα αποστείλει εκ μέρους της Γαλλικής Γερουσίας είχαμε κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Παρατηρήσαμε ότι οι παρατηρήσεις αυτές αποτυπώνονται ορθώς στο τελικό κείμενο σύνθεσης. Αυτό είναι ένα θετικό σημείο το οποίο υπόσχεται καλά για τη συνέχεια. Να δώσω τώρα κάποιες πληροφορίες σχετικά με την Γαλλική Δημοκρατία και με τις εξελίξεις της επόμενες εβδομάδες. Η Επιτροπή μας Οικονομικών Υποθέσεων ασχολείται με δύο βασικά κείμενα, στα οποία θα υπάρξουν εκθέσεις. Από τη μία υπάρχει η διαδικασία επικύρωσης και από την άλλη υπάρχει ο οργανικός νόμος για την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν τα δημοσιονομικά στη χώρα μου. Όπως γνωρίζετε όλοι, είναι προφανές ότι το σύμφωνο θα επικυρωθεί από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, δηλαδή στην Γερουσία η παρούσα αριστερή πλειοψηφία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε αφεαυτής να επικυρώσει την διαδικασία εάν οι ψήφοι της αντιπολίτευσης δεν ακολουθούσαν. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, γιατί αυτό στην ουσία δίδει θα έλεγα ε, μια ευρεία πολιτική βάση. Μετά ο οργανικός νόμος. Σε επίπεδο γαλλικού δικαίου είναι το επίπεδο το άμεσα κατώτερο από τον συνταγματικό χάρτη. Ο οργανικός αυτός νόμος θα καθορίσει με συγκεκριμένο τρόπο τις λεπτομέρειες θα αναφέρεται στα στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν τη σύγκριση των δημοσιονομικών εγγράφων των χωρών της ζώνης ευρώ και ο οργανικός αυτός νόμος για πρώτη φορά στη Γαλλία θα δημιουργήσει αυτό το οποίο οι οικονομολόγοι ονομάζουν ανεξάρτητη δημοσιονομική επιτροπή, μια επιτροπή εμπειρογνωμοσύνης και παρακολούθησης των εξελίξεων. Αυτό το συμβούλιο λοιπόν το Ανώτατο Συμβούλιο θα έχει ένα ουσιαστικό ρόλο για να εγκρίνει τις μακροοικονομικές ε, προβλέψεις, για να αναπτύσσει σταδιακά έννοιες όπως ο οικονομικός κύκλος, διαρθρωτικό έλλειμμα, διαρθρωτικές προσπάθειες, έννοιες σχετικά με τις οποίες οι δράσεις των μεν και των δε οφείλουν να τίνουν προς το 3% και την πορεία επιστροφή στην ισορροπία στα πλαίσια της πολυμερούς παρακολούθησης, εποπτείας. Λοιπόν, Πρόεδρε, συμφωνώ με την συνέχιση αυτής της ευρωπαϊκής απόπειρας και, Πρόεδρε, θα ήθελα σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιμένω στο τακτά χρονικά διαστήματα, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία κάποια συμφωνία. Οι προσανατολιστικές γενικές συζητήσεις πάντα παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον βέβαια, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον, στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας, θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα, έτσι ώστε με μεθοδικό τρόπο να εμβαθύνουμε αμοιβαία στην γνώση των προσπαθειών του καθενός. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μπάουλς ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιονομικών της Βελγικής Γερουσίας, ο κύριος Ζιλκινέ. Έχετε το λόγο κύριε Ζιλκινέ για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία στην παρούσα φάση να ενισχύσουμε τον διάλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Θα προχωρήσω άμεσα στις συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Από τη μία είμαστε υπέρ της διαδικασίας, ε, ε, θα έλεγα, ελέγχου των δημοσιονομικών. Από την άλλη έχουμε, θα έλεγα, στις συστάσεις προς το Βέλγιο κάποιες αντιρρήσεις. Τέσσερις αντιρρήσεις. Καταρχάς, περιορίζεται η προσοχή στην, στον περιορισμό των δαπανών αγνοώντας τα νέα έσοδα σε σχέση με τον φόρο για τις ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες κτλ. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα και στην πολιτική ανάκαμψης και στην πολιτική που προστατεύει ε, ε, τα κοινωνικά συστήματα προστασίας και εσείς ξέρετε ότι εμείς εμένουμε στο Βέλγιο στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αμοιβών, των μισθών. Δεύτερον, ξεχνάμε ορισμένες σημαντικές διαστάσεις τη διαδικασία 2020, τους δείκτες για την καταπολέμηση της ένδυας, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη, των κενών και ελλείψεων στον τομέα της ενέργειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αγνοούνται και δεν μπορούν να αγνοηθούν αν θέλουμε να προετοιμάσουμε τις θέσεις εργασίας και την οικονομία του αύριο τρίτο στοιχείο είναι η ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μέσα σε έναν επαναπροσανατολισμό της οικονομίας, υπέρ της πραγματικής οικονομίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικολογική μεταβατική φάση της οικονομίας, κάτι το οποίο σύμφωνα με πολλές εκθέσεις είναι πηγή θέσεων εργασίας για το μέλλον. Και τέταρτον, ε, δεν δίδεται η απαιτούμενη προσοχή στην μεταρρύθμιση του πιστοτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, κάτι το οποίο προκάλεσε όπως ξέρετε ένα μεγάλο τμήμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη σήμερα. Και στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη, περισσότερη πολιτική βούληση σε σχέση με τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών ε, δραστηριοτήτων πράξεων. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές, τον εισηγητή για το σχέδιο το οποίο μας καταθέτει σήμερα θα πρέπει να εξελιχθεί συμπεριλαμβάνοντας και θέματα φορολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά έτσι ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη συνένεση θα πρέπει στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχία να προσθέσουμε και τις διαστάσεις αυτές που ανέφεραν θέλουμε να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ κύριε Ζελκίνε. Την Έμιλι Τέρμαν έχει το λόγο. Όχι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι. Εγώ είμαι από τους Πράσινους ε, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο από τη Δανία που παρακολουθούμε το εξάμεινο ακόμα και αν δεν είμαστε στο Ευρωζώνη όπως είπε και ο Σουηδός εκπρόσωπος. Εμείς ε, Θεωρούμε πως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να συζητηθούν οι ανισορροπίες, να μειωθεί, να δούμε ποια είναι η πίεση που ασκείται και να έχουμε μια κοινή ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση καθώς και τη δυνατότητα συντονισμού, κάτι το οποίο θα μπορούσε και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Το υποστηρίζουμε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και χώρος για βελτίωση σε σχέση με το τι ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να βρούμε σωστή ισορροπία ανάμεσα στους οικονομικούς στόχους και τους στόχους 2020 ε, ε, πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα και έπειτα να υπάρξει μια συνοχή ανάμεσα στα δύο αυτά που για την ώρα φαίνεται να είναι αντιφατικά κάποιες στιγμές, ενώ δεν θα έπρεπε. Επίσης μας ε, προβληματίζει το αν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε, να παρακολουθήσουμε από τα πρώτα έτη εφαρμογής ε, το τι εφαρμόζεται και τι όχι. Ε, και να μην προχωράμε έτσι στα τυφλά, να έχουμε πραγματικές συστάσεις και οι προτεραιότητες ε, της ε, κυβέρνησής μου επαναλήφθησαν σε κάποιο βαθμό και ίσως κάποιες φορές θα έπρεπε να αμφισβητώνται όλα αυτά λίγο περισσότερο. Και μια τελευταία παρατήρηση είναι, όπως αναφέρθηκε, είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, που πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό σημείο, ιδιαίτερα σε σχέση με τους στόχους του 2020, είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσά από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζω πως ε, και εσείς ε, θα μας πείτε ποια θεωρείτε ότι είναι τα ωφέλη αυτού του εξαμήνου και ποια μπορεί να είναι τα δυνητικά προβλήματα επί των οποίων θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε το εξάμεινο πραγματικά να λειτουργήσει και να ωφελήσει. Σας ευχαριστώ. Πώ λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ε, τώρα οι επόμενοι δύο εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, ο Άλεξ Γουάιτ, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για τις Δημόσιες Δαπάνες και τις Μεταρρυθμίσεις, και έπειτα ο, Ολγκράντο Καμπίτα από την Πορτογαλία, επίσης επικεφαλής της Επιτροπής για τον Προπολογισμό και την Οικονομία. Έχεις το λόγο, Άλεξ. Αν δεν ξέρεις που είναι τα κουμπάκια για τα μικρόφωνα, είναι μπροστά σα και ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή απόψε ε, και την δυνατότητα επαφής ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια, τους Εθνικούς Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές σε σχέση με την προσέγγιση αυτή του εξαμήνου, την οποία καλωσορίζω, νομίζω πως είναι σημαντικό σημείο εκκίνησης για όλους μας για όλους όσους έχουμε ένα πρόγραμμα ας πούμε, που μας ε, οδηγεί κατά τη διάρκεια του ναι. έτους για το πώς διαχειριζόμαστε από κοινού την ευρωπαϊκή διάσταση των όσων πρέπει να κάνουμε ώστε να προοδεύσουμε μετά και από το εθνικό εξάμεινο. Να πω δύο λόγια για την Ιρλανδία και ίσως να επανέλθω σε γενικότερα ζητήματα όπως τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Η Ιρλανδία είναι σε πρόγραμμα βοήθειας και ε, προχωράμε, προοδεύουμε και σε συνδυασμό με όλες αυτές τις πτυχές ε, που έχουμε ήδη συμφωνήσει, το Κοινοβούλιο και η δική μου Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, σε σχέση για παράδειγμα με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την πολιτική για την αγορά εργασίας, ε, την πολιτική για τις συντάξεις. Υπάρχουν κάποιες, ε, ε, κάποια προβλήματα τα οποία χρειάστηκε να τα αντιμετωπίσουμε ως Επιτροπή και όσον αφορά αυστηρά την, επιτροπή, την εφαρμογή του ίδιου του εξαμήνου και των συστάσεων, θα με ενδιαφέρει να ακούσω από συναδέλφους από άλλες χώρες πώς προχώρησε, γιατί εμείς είμαστε σε ένα πρόγραμμα βοήθειας, υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός ελέγχου. Πολλοί θα έλεγαν ότι υπάρχει και μεγάλη παρέμβαση και εμπλοκή της Τρόικα στη διαχείριση των, της οικονομίας μας. Ε, η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο όμως κατάφερε να μείνει, ε, να συμβαδίσει με τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούν την ε, Ιρλανδική κοινή γνώμη αλλά το πλαίσιο αυτής της βοήθειας είναι ασύνηθες πλαίσιο για οποιαδήποτε χώρα και έχει αντίκτυπο στην φύση, στο επίπεδο και την, ε, της δημόσιας συζήτησης. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κάνουμε ωστόσο ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε ενήμεροι και διαρκώ ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Το εξάμενο είναι σημαντικό και θα είναι σημαντικό και στο μέλλον και ίσω να μπορέσουμε πιο στενά ακόμα να το εφαρμόσουμε καθώ θα προχωράμε και καθώ θα βγούμε από το πρόγραμμα βοήθεια όπω αναμένουμε ε, σύντομα. Να πούμε και πάλι ότι είναι σημαντική αυτή η διαδικασία για μας και ίσως θα πρέπει να γίνει συζήτηση, ίσως όχι σήμερα, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την ισορροπία ανάμεσα στο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί έχουμε χωριστές ε, ε, αρμοδιότητες αλλά και επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος. Πρέπει κάπως περισσότερο λοιπόν να το σκεφτούμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει το άρθρο 13 της, ε, του Συμφώνου Σταθερότητας. Ε, θα ήταν ευπρόσδεκτη μια τέτοια ευκαιρία για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ε, να επιβεβαιώσω ότι όντως θα εξετάζουμε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρατε, γιατί είναι κάτι που όντως θα πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί δεν μπορούμε όλη την ώρα να σας τραβολογάμε εδώ. Από την Πορτογαλία, ο κύριος Καμπρίτα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και οι επιτροπές που εδώ αντιπροσωπεύονται σήμερα, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διάλογο για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, γιατί ε, έτσι έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε αυτή τη φάση της κρίσης, όπου η ταυτότητα του ευρωπαϊκού ε, οράματος αμφισβητείται σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία, η οποία είναι σε μια διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική ε, και διαδικασία προσαρμογής είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη στην αξία του ευρωπαϊκού οράματος και είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι συμμετοχικές διαδικασίες και είναι τα κοινοβούλια που είναι η φωνή των λαών και αντιστοιχούν σε ένα όραμα μιας Ευρώπας απαιτητικής αλλά αλληλέγγυας και δημοκρατικής και αυτό απαιτεί περισσότερο διάλογο και συμμετοχή των κοινοβουλίων. Η Πορτογαλία ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανάπτυξης διαδικασιών πολιετούς προγραμματισμού οικονομικού με τη θέσπιση στόχων δαπανών ε, τετραετία, που ξεκίνησαν άρχισαν μάλλον να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έγιναν εδώ και δύο χρόνια πρέπει να ολοκληρώσουμε και να ενσωματώσουμε και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και έχουμε και τις ειδικέ απαιτήσει μιας χώρας η οποία όπως ξέρουμε ε, ισχύει το μνημόνιο για διεθνή βοήθεια. Σε αυτό το πλαίσιο η Πορτογαλία έχει μια αντίληψη για τη δημόσια οικονομία ανεξάρτητη. Έχουμε, τρεις, ε, έχουμε μια επιτροπή όπου συμμετέχουν ε, τρεις Πορτογάλοι και δύο που συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως είναι αποφασιστική σημασία να δεσμευτεί η προσπάθεια μάλλον να συνδυαστεί η προσπάθεια δημοσιονομικής πειθαρχίας με ένα όραμα συγκεκριμένων στόχων ε, ανταγωνιστικότητας μέχρι το 2020 και άρα με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Πορτογαλία, στην Πορτογαλία υπήρξε συνένεση για όλα τα μέτρα μεταρρύθμισης, αλλά θα πρέπει να πω εδώ με μεγάλη ανησυχία πως βλέπουμε πως στην πράξη το πρόγραμμα προσαρμογής ε, οδήγησε σε τεράστια αύξηση της ανεργίας από το 12% στο 16% τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο, ψηλότερο ποσοστό που έχουμε ποτέ φτάσει και έχουμε φτάσει σε επίπεδα ύφεσης πολύ πιο πάνω από αυτά που αρχικά προβλέπονταν από το πρόγραμμα. Και γι' αυτό σε αυτή την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συνδυάσουμε συντονισμό των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας με ένα όραμα που επιτρέπει να δημιουργείται μια, μάλλον να υπάρχει προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο και στο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία των προσαρμοστικών προγραμματωμάτων. Το, το εξαπλό μέτρο και το διπλό μέτρο θα πρέπει να συνδυάσουν αυτή την, αυτά τα μέτρα ε, αύξηση της αντιγωνιστικότητας αλλά και της ε, αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, εξ ε, της ομάδας ECR, ο κύριος Έπινγκ στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές παρατηρήσεις για τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα της άσκησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, πρέπει να πω ότι συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά λίγα μόνο νέα έχει να προσφέρει και ο ΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο για χρόνια, για να μην πω δεκαετίε, τι ίδιε συστάσει κάνουν. Και πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στα κράτη-μέλη να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία ήδη πράττουν. Και όπου αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη-μέλη τείνουν να αγνοούν τι συστάσει ή να κάνουν το ακριβώ αντίθετο. Ηπό την έννοια αυτή, 1.500 σελίδε αναλύσεων και κατευθυντήριο γραμμών πολιτική φαίνονται λίγο άσκοπε. Η να κανουν το ακριβω αντιθετο υπο την εννοια αυτη 1500 σελιδε αναλυσεων και κατευθυντηριου γραμμων πολιτικη φαινονται λιγο ασκοπε η γαλλια θα δεχτεί διαταγές από τις Βρυξέλλες υπαριθμών ένα σύσταση για τη Γαλλία είναι να δουλεύει ο κόσμος περισσότερο και όχι λιγότερο. Το πρώτο πράγμα όμως που ο κύριος Ολάντ έκανε και μου αρέσει το όνομά του γιατί είμαι Ολλανδός είναι να μειώσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Και είναι αμφίβολο αν θα συνεχίσει τη λιτότητα που του συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο κάτω-κάτω εξελέγει με υποσχέσεις τελείως κατά της λιτότητας. Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό διάλογο που ε, μας αφορά εμάς, θα ήθελα να θυμίσω εδώ στην Επιτροπή την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με τον Υπουργό Οικονομικό του Βελγίου, τον κύριο Βανάκερε. Ε, πολύ ρόδινα μας τα περιέγραψε τα θέματα της βελγικής οικονομίας. Και τώρα φαίνεται ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η παρουσίασή του ήταν υπεραισιόδοξα. Αντί να είναι Υπαριθμόν ένα στις επιδόσεις το Βέλγιο οδεύει προς την ύφεση. Συρρυκνώνεται η οικονομία με υψηλότερους ε, ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά φάρσα ήταν αυτό που είδαμε ε, για όλη διαδικασία και ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Δεκρό, ε, πρώην πρόεδρος της Βελγικής Βουλής, θα συμφωνήσει και το καλωσορίζω κατά τα άλλα ενώπιόν μας. Ο οικονομικός διάλογος με το Βέλγιο βασικά δεν είπε ε, δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα ωραίο σοου για τον χώριο τύπο. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή μας ήταν μάλλον περιορισμένη. Επίσης, αυτό φάνηκε και από τη χαμηλή το προσέλευση των μη Βέλγων βουλευτών. Βασικά ήταν ένας Βέλγος υπουργό και κυρίως Βέλγοι ευρωβουλευτές ε, στο διάλογο αυτό. Και πιο σημαντικό ακόμα, είναι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την ευέλικτη αγορά εργασίας, ε, αηφόρα, συνταξιοδοτικά συστήματα και βιώσιμα και μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους επόμενους δύο εκπροσώπους Εθνικών Κοινοβουλίων από τη Λετωνία, τον Γιάννη Σοζολίνης, και από τη Λιθουανία ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ο κύριος Καστρούζης. Right. Mr. wherever you are. Ο κύριος Οζορίνης έχει το λόγο, δεν ξέρω που βρίσκεστε, από τη Λετωνία. Ελπίζω να καταλάβατε ε, ότι σας εννοούσα. Ναι, το όνομα της χώρας μου το είπατε καλά, λέει ο εκπρόσωπος της Λετωνίας. Για να με καταλάβετε θα ομιλήσω τη λετονική. Συμφωνούμε λοιπόν με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουν γίνει οι απαιτούμενες συζητήσεις με το Συμβούλιο και τους εκπροσώπους της Επιτροπής θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία των αποτελεσμάτων από τα έγγραφα του ε, εξαμήνου. Απαιτείται να βελτιώσουμε επίσης και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αν θέλουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Νομίζω πάντως ότι το πρόγραμμα αυτό της σύγκλησης και τα εθνικά προγράμματα μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα καθιστώντας μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εφικ... καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εφικτό έχοντας βέβαια ανάγκη ε, κάποιας, κάποιους μακροοικονομικούς δείκτες τα μεταρρυθμιστικά εθνικά προγράμματα θα πρέπει να ελέγχονται μεν σωστά. Ε, νομίζω ότι θα είχαμε ε, καλύτερη γνώση της κατάστασης αν ήταν τα στοιχεία πιο αξιόπιστα. Επιπλέον χρειαζόμαστε ε, περισσότερες ε, πληροφορίες από τις έκτακτες συνεδριάσεις των Συμβουλίων. Και στην αρχή ε, υπάρχει περισσότερη δουλειά, γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός και οργάνωση σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σύγκλησης και τα εθνικά σχέδια. Για τη Λετωνία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η δυνατότητα, να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δυνατότητα, να φέρνει διευκρινήσεις ε, για τις συστάσεις. Μπορεί να μην αλλάξουν οι συστάσεις στην ουσία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγκαίρως να κάνει σχόλια η χώρα ε, για να ε, μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Παράδειγμα, για το 2012, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαλόγου, έτσι να είναι διπλής κατεύθυνσης αυτή η υπόθεση. Επίσης, ε, οι ημερομηνίε ε, θα πρέπει να είναι πιο ελαστικές, όχι τόσο απόλυτα τα χρονικά περιθώρια. Επίσης, συμφωνεί η Λετωνιώτη στα πλαίσια ε, του εξαμήνου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης των επίκαιρων θεμάτων και επιγόντων που δεν λύνονται στο Συμβούλιο. Παράδειγμα, η δημοσιονομική πολιτική. Αυτό θα βοηθούσε να μην γίνονται διπλές συζητήσεις και επικαλύψεις και παράλληλα, να γίνονται εγκαίρως παντού και ε, επίσης το ευρωπαϊκό εξάμεινο να είναι απλό και με διαφάνεια και οι φυστάμενες πρωτοβουλίες να μην υπονομεύονται ή να μην πολλαπλασιάζονται. Ευχαριστώ. Lithuanian Committee on Budget and Finance, Mr. Και τώρα ο κ. Γκλαβέτη από το Λιθενικό Κοινοβούλιο, πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Προπολογισμού και Οικονομία. Σα ευχαριστώ. Πολύ προλαλήσαντες όρισαν ε, και περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα, ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Στη Λιθουανία λέμε ότι δεν μπορούμε να τα μπερδεύουμε και να τα αναμειγνύουμε όλα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές εθνικές καταστάσεις. Όπως και άλλες χώρες, η Λιθουανία αντιμετωπίζει την κρίση και η κυβέρνηση καθώς και το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας έλαβε διάφορες επιτυχείς αποφάσεις. Πρέπει να, παραδεχτούμε ότι είχαμε αρκετή επιτυχία ε, γιατί αξιολογήσαμε τα διδάγματα που, είχαμε αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι προβλέψεις για φέτος και του χρόνου δείχνουν ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 3% ε, έλλειμμα. Οι μεταρρυθμίσεις επίσης εφαρμόστηκαν αρκετά επιτυχώς. Αφού ακούσαμε τι, όσα είπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω πως κατά τη γνώμη μας το εξάμεινο, το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ σημαντικό ψυχολογικά. Στη Λιθουανία, στη Λιθουανία παρατηρήσαμε ότι πολλές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη δημόσια οικονομία, τα κοινωνικά συστήματα πρόνοιας, ε, έχουν να κάνουν όχι μόνο με την, τα οικονομικά ζητήματα, αλλά με ψυχολογικά ζητήματα. Για παράδειγμα, το Λιθωνικό Κοινοβούλιο προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για τις εκλογές. Ο νέος προϋπολογισμός θα υιοθετηθεί από το νέο κοινοβούλιο και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις γενικές αρχές, την ε, δημοσιονομική πολιτική και η ευρωπαϊκή στήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική για μας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω πως οι συζητήσεις ε, είναι εξαιρετικά σημαντικές όταν έχουμε να κάνουμε με την ε, ψυχολογική πτυχή της κρίσης. Εν τέλει θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμενο είναι ένας τρόπος για αναζήτηση λύσεων στη δημόσια οικονομία, στα, στα δημοσιονομικά στα θέματα, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις και στον ψυχολογικό τομέα και νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να είναι πρόσδεκτος προς αυτή την άποψη. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε χρόνο μάλλον για μία-δύο ερωτήσεις επιπλέον από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν κανείς κρατιέται και δεν έχει ζητήσει το λόγο, μπορεί να το κάνει. Τώρα εξ των Πρασίνων, ε, όχι συγγνώμη, από την εξονόματος της Γκουε, η Μαρίζα Ματίας. Όχι, δεν άλλαξε ακόμα ομάδα, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Όπως και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από λίγο, Θα ήθελα όλους να σας καλωσορίσω για αυτή τη συζήτηση, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική και θα ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια σε σχέση με την θέση του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα. Καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Γκοζές για την πρόταση που έκανε και για την απόπειρα συμφιλιασμού, συμφιλίωσης μάλλον διαφορετικών απόψεων στο θέμα και κυρίως αξιοποίησης αυτού που φαίνεται να είναι και εκτιμένο στη συζήτηση που κάνουμε, δηλαδή αυτή την προσπάθεια εξισορρόπησης των μηχανισμών δημοσιονομικής πειθαρχίας με τους στόχους ανάπτυξης που είναι ε, θεμελιώδης σημασία. Η δουλειά που κάνατε προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνει. Δηλαδή οι πολιτικές και η πραγματικότητα που ζούμε είναι πολλές φορές ε, ε, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή οι πολιτικές που ασκούνται δεν ε, οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρέπει ε, ωστόσο να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ε, Ποια είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Αυτό είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η ανεργία, η έλλειψη ανάπτυξη. Έχουμε προβλήματα πολύ διαφορετικά, σε πολύ διαφορετικέ καταστάσει στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν μόνο ένα ομοιόμορφο μέτρο. Χρειάζονται απελπιστικά, χρειαζόμαστε λύσει από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία ε, που ε, ε, επίση βρίσκεται υπό καθεστώ η δημοσιονομική πειθαρχία τη σημαίνει λιτότητα. Αυτό είναι το συνώνυμο. Δηλαδή δεν μιλάμε καθόλου ούτε για δημόσιες επενδύσεις, ούτε για δημιουργία απασχόληση. Τα όσα λέμε για συντονισμό τελικά ε, σημαίνει πειθαρχία, λιτότητα των χωρών του Νότου ε, για να επιτύχουν κάποιους στόχους. Ενώ όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό όραμα θα πρέπει να έχουμε ισότητα ευκαιριών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την ε, μανία, την αιμονή της ε, κάλυψης του χρέους. Βρισκόμαστε σε κρίση στην Ευρώπη με τελμάτωση και ύφεση σε πολλές ε, περιφέρειες. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής είναι μέτρα δημοσιονομικού τύπου, ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, η ευελιξία ε, των, στα, στα εργατικά δικαιώματα ε, και στην Πορτογαλία και στις υπόλοιπες χώρες είναι όλα αυτά πολύ, πολύ ορατά. Πρέπει ωστόσο να προσπαθήσουμε να βρούμε καλύτερη συνοχή και σύγκληση των οικονομιών, όχι με, τον τρόπο μόνο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ένα κοινό πρόγραμμα που να μην τιμωρεί τους νότιους. Ε, χωρίς καμιά αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουμε από το Λουξεμβούργο τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, τον κύριο Ροζέ Νεγκρή και από το Βελγικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Ντεκρούν. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε λοιπόν για την εισαγωγή που κάνατε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στον προϋπολογισμό από τη μία και την δημοσιονομική πειθαρχία και από την άλλη την ανάγκη να ξεκινήσει η οικονομία να δουλεύει πάλι και μέσω των δημοσίων επενδύσεων και μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Αναφερθήκατε σε θέματα όπως η ανεργία των νέων, προβλήματα ή σε θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών. Ε, τα προβλήματα αυτά δεν έχουν ακόμα λυθεί. Έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά στη χώρα μας, όπως το σύστημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, που όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν αποδείξει την αξία τους. Αυτό το οποίο επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι σε ποιο βαθμό τα κράτη της Ευρώπης, τα, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να σημειώσουν βήματα προόδου και να βοηθήσουν και άλλες χώρες να διατηρήσουν την δημοσιονομική και πολιτική τους ανεξαρτησία. Θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να είναι ένα σύστημα ε, ζωντανό το οποίο να βελτιώνεται συνεχώς και είναι απαραίτητο να είμαστε βέβαιοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια των κρατών μελών θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα, μια κατάσταση θα έλεγα διαδοχικών αξιολογήσεων, παρακολούθησης των μέτρων που έχουν αποφασιστεί και εφαρμόζονται και αξιολόγησής τους. Πιστεύουμε ότι έτσι ε, ε, θα μπορούμε να κάνουμε και νέες συστάσεις εφόσον αυτό είναι το απαραίτητο. Διατηρώντας την εθνική μας αυτονομία βέβαια. Ο κύριος Σερμάντο Κρού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας εκπλήξω λίγο λέγοντας ότι είμαι μέλος του κοινοβουλίου μου για 44 χρόνια. Από το 68 μέχρι σήμερα έχω αναλάβει διάφορες θέσεις και σε αυτά τα 44 χρόνια έχω δει την μάχη θα έλεγα ανάμεσα στον, ε, σε αυτούς που είναι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και σε αυτούς οι οποίοι α, χάνουν την εθνική κυριαρχία και το διαπιστώνουν αυτό. Ε, υπήρξαν ε, τέτοια φαινόμενα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, φαινόμενα τα οποία έχουν ε, από τη μία αναπτύξει τις αγορές, έχουν βοηθήσει την οικονομία και έχουν κατά κάποιο τρόπο ισορροπήσει τα θέματα του ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών γενικότερα. Βέβαια αυτό δεν ίσχυσε για όλες τις χώρες. Πολλές χώρες κράτησαν μια πολιτική θα έλεγα εθνικά κυρίαρχη υπεύθυνη και δημοκρατική απέναντι στους, στο εκλογικό του σώμα. Μέχρι τη στιγμή βέβαια που είδαμε μπροστά μας την κρίση, οπότε διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να είχαμε την πολιτική ένωση αν δεν είχαμε ορισμένα κριτήρια αντιστοιχίας στα πλαίσια της λειτουργίας της οικονομίας. Και αρχίσαμε λοιπόν να συζητάμε με βάση άλλα κριτήρια πλέον, όχι εθνικής κυριαρχίας, αλλά ελίματος δημοσίου χρέους, αξίας των νομισμάτων. Και αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη και στη δική μου χώρα και στην Ισπανία και αλλού, είναι καταστάσεις ε, έκτακτες και η προσαρμογή των χωρών ε, με τρόπο θα έλεγα που δείχνει τη στροφή τους προς το έσω ε, είναι κάτι το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Δεν χρειάζεται για να συνδυάσει κανείς την δημοσιονομική ορθοδοξία και την ανάκαμψη να λειτουργήσει με εσωστρέφεια σαν χώρα. Αν η Ευρώπη είχε το θάρρος και τα μέσα να προχωρήσει στην οικονομική ανάκαμψη, σεβόμενη την δημοσιονομική πειθαρχία και ορθοδοξία, είμαι βέβαιος ότι θα είχαμε κάνει τα απαιτούμενα βήματα. Τη απουσία ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα είναι τώρα στην διεθνή σκηνή τα 47 χρόνια που είμαι κοινοβουλευτικός είδαμε τι έγινε με την Κίνα, με την Ινδία, με την Ινδονησία, με τη Βραζιλία. Είναι χώρες ανταγωνιστικές με τεράστιες ικανότητες που έφεσαν πλέον σε αμφισβήτηση το σύστημα με το οποίο κινηθήκαμε μέχρι τα τελευταία χρόνια. Να λοιπόν η συζήτηση που γίνεται ε, είναι μια συζήτηση που έχει σχέση με το πώς θα αντιμετωπίσει κάθε χώρα με εσωστρέφεια ή όχι το πρόβλημα και πώς θα προχωρήσει στην ανάκαμψη. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητές από πλευράς της Επιτροπής, η κυρία Μπερές πρώτα και πως θα προχωρησει στην ανακαμψη ευχαριστω δυο ομιλητες απο πλευρα της επιτροπης η κυρια μπερετς πρωτα και μετα ο Σφεν Γκίγκολτ. Και μετά θα επανέλθω στον εισήγητη. Εκτός αν κάποιος άλλος ζητήσει το μεταξύ το λόγο υπερβάνς. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίδεται να συζητήσουμε με ορισμένους εκπροσώπους κοινοβουλίων των κρατών μελών την διαδικασία που εκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσει η κρίση. Και βλέπουμε τι σημασία έχει αυτή η διαδικασία. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, εμείς και τα κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού αν θέλουμε πράγματι να έχουμε πίστη όχι στο υπερπέραν αλλά στην αποτελεσματικότητα του εξαμήνου μας. Σε επίπεδο Συμβουλίου υπάρχει κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Στην ουσία βρισκόμαστε ακόμα στα δύσκολα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, έχουμε εξέταση των προτάσεων, έχουμε την πρόταση για την εξέταση των εθνικών σταθεροποιητικών προγραμμάτων και τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά γενικοί προσανατολισμοί από πλευρά στο Συμβούλιο, βλέπουμε ότι έχουμε ειδικέ συστάσεις από χώρες, για χώρες συγγνώμη, συγκεκριμένες. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν εδώ κάποια διφορούμενα στοιχεία, δημιουργικής φαντασίας ίσως, αλλά τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν. Ο εισηγητής εξέφρασε απέναντι στα κοινοβούλια των κρατών μελών τις ιδέες του για το πώς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους εν αρμονία. Ε, Από αυτή την άποψη η πρώτη μελέτη την οποία κάναμε το πρώτο τμήμα μάλλον της μελέτης την οποία κάναμε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μου είχε φανεί λίγο απογοητευτική. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε τώρα μπροστά μας είναι μια χρησιμότατη βάση. Γιατί πραγματικά είναι μια εξέταση εκ των κάτω προς τα άνω για τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τα θέματα τα οικονομικά τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Για να με καταλάβετε θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου γιατί στη σελίδα 15 όπου υπάρχει μια απλουστευμένη θα έλεγα παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπάρχει μια κενή γραμμή, μια κενή ρήγα που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι γιατί είμαστε άχρηστοι εμείς, αλλά αν θυμάμαι καλά, από το 2004 διοργανώνουμε συναντήσεις με τα κοινοβούλια των κρατών μελών για να επηρεάσουμε ακριβώς το Συμβούλιο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι κάνοντας το αυτό, συνεχώς ε, θα έλεγα τροπολογούμε με τον τρόπο μας τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να διαβάσουν πάρα πολύ προσεκτικά τα συμπεράσματα της μελέτης αυτές για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι πολύ αποτελεσματικές οι προτάσεις αυτές γιατί βασίζονται ακριβώς σε μια σωστή ανάγνωση των προηγούμενης εμπειρίας, της προηγούμενης εμπειρίας. Να πούμε ότι στα πλαίσια της Επιτροπής μας έχουμε βοηθήσει και εμείς στη σύνταξη της εκθέσεως Γκοζές με δύο τρόπους. Δηλαδή πρώτον, Υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κανονικά τα κράτη-μέλη θέτουν στην τράπεζα των συζητήσεων τα εθνικά τους προγράμματα για την απασχόληση. Κάποιες χώρες το έκαναν, κάποιες άλλες δεν το έκαναν και σκοτίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν το έκαναν. Ε, αυτό δεν είναι καθόλου καλό γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες που δούλεψαν καλά δεν είχαν λόγο να δουλέψουν και αυτές οι οποίες δεν δούλεψαν δεν τους έγινε και καμία παρατήρηση. Είμαστε σοβαροί λοιπόν και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να ελέγχει το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη ή κάνουμε πράγματα που δεν έχουν νόημα. Πρέπει λοιπόν για τον επόμενο χρόνο και η μεν και η δεν να εξηγήσουμε τι περιμένουμε για τα προγράμματα ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των κρατών μελών και την αδυναμία τήρησης του χρονοδιαγράμματος στο σύνολο της Ευρωζώνης και από την άλλη να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα οποία κάνει και συστήνει η μία χώρα επηρεάζει και τις άλλες χώρες. Υπάρχει το λεγόμενο φαινόμενο spillover που ε, μεταδίδεται το πρόβλημα μίας χώρας πολύ εύκολα πλέον στις υπόλοιπε. Σας άφησα να συνεχίσετε γιατί δεν πιεζόμαστε και τόσο πολύ χρονικά. Τελευταίος ομιλητής είναι, ομιλητής είναι ο Σφεν Γκίγκολντ. Θα Ήθελα απλώς να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι χρήσιμη. Πρώτον, για αυτό που είπε η Περβάνς. Όταν πληρώνουμε για μελέτες, καλό είναι να τους ζητούμε να μας συμπεριλαμβάνουν και εμάς. <laughs> Θα το συζητήσουμε με τους φίλους μας του Μπρόγγελς ε, κατά τα άλλα, έτσι λίγο πιο σοβαρά, ε, νομίζω ότι το πρόβλημα τώρα που διαπιστώνουμε με τη διαδικασία αυτή είναι ότι πολλές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κατά την άποψή μου αρκετά χρήσιμες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα διότι κάποια ζητήματα της στρατηγικής Ευρώπης 2020 δεν συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο επίπεδο με κάποια άλλα και θα πρέπει να επιμένουμε περισσότερο. Ας πούμε, η καταπολέμηση της ένδυας ε, ή ζητήματα στόχων περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών θα πρέπει να τονιστούν περισσότερο. Αλλά πολλές από τις συγκεκριμένες ε, συστάσεις, αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου φαίνονται λογικά και χρήσιμα ε, για τις χώρες που εγώ γνωρίζω περισσότερο και ιδιαίτερα για τη Γερμανία. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, ότι πολύ συχνά Κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται οι ίδιες συστάσεις και οι περσινές είναι ίδιες με τις φετινές. Και προσβλέπω και σε μελλοντική ανταλλαγή απόψεων μαζί σας να μου πείτε πώς το βλέπετε. Γιατί για τη Γερμανία όλες οι βασικές συστάσεις είναι πανομοιότυπες, διότι δεν άλλαξε απολύτως τίποτα στην ουσία. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απουσιάζει τώρα και μάλλον δεν τολμάει να το πει ξεκάθαρα. Ας πούμε, Ε, υπάρχουν ε, συστάσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην παιδεία άτομα με αναπηρίες. Ωραία, κάτι άλλαξε, μπορεί να είναι περιφερειακές αλλαγές, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλες. Το ίδιο ισχύει ε, και με τον υψηλότερο φορολογικό συνδελεστή ε, ορισμένοι άνθρωποι που είναι εύποροι και έχουν μεγάλη περιουσία δεν τους συμφέρει να εργάζονται γιατί τους θα παίρνει εφορία. Λοιπόν, ε, εσείς πώς αξιολογείτε ε, συγκεκριμένα τις διάφορες προτάσεις, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και αυτή είναι πραγματικά η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Μου άρεσε πολύ ε, παρατήρηση του συναδέλφου της Γαλλικής Γερουσίας που είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τα διάφορα θέματα γιατί εκεί γίνεται η ουσιαστική συζήτηση και όχι αφηρημένη. Αυτό χρειαζόμαστε έτσι ώστε να ε, ε, λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό εξαμένο. Λοιπόν, ας κάνει ο καθένας τα μαθήματά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να είναι πιο ε, αυστηρή και μεγαλύτερη διαφάνεια ποιος ανταποκρίθηκε και ποιος όχι και να μην τα κρύβουν αυτά κάτω από διάφορα έγγραφα εργασία ή μέσα σε έγγραφα εργασία. Ε, να συζητούμε σε μεγαλύτερο βάθος τα διάφορα ζητήματα και τότε και σε σύγκριση με τη στατική της Λισαβόνας ε, αυτό συνιστά πραγματική πρόοδο και πρόοδο που μας χρειάζεται οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή μας. Δεν ξέρω θέλει κανένας άλλος να μιλήσει. Παρακαλώ, Ζαν Πολ Γκοζέσν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις παρεμβάσεις όλων και ιδιαίτερα των συναδέλφων μας ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι σε αυτή την άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις διευκρινήσεις που κάνουμε τώρα με διαδοχικές εκθέσεις, αυτό που έχει σημασία είναι να διασκεδαστούν ορισμένοι φόβοι. Άκουσα να λέγουν αρκετοί ότι στις χώρες τους υπάρχουν ιδιαιτερότητες τις οποίες ε, θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη και να φροντίσουμε να μην ε, διακυβευθούν. Ας πούμε, για το πόσο ορίζονται οι μισθοί, ε, όπως ανέφερε ο Σουηδός συνάδελφος. Κάτι άλλο που είπε ο συνάδελφος από την Αυστρία είναι ότι μακροπρόθεσμα ε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα, γιατί ε, στην Αυστρία είναι πολυετής αυτή η άσκηση, αλλά δεν μπορεί το ευρωπαϊκό εξάμεινο να ε, αναχθεί σε μια παρακολούθηση και μόνο. Πρέπει να είναι μια δυναμική διαδικασία, να κάνει και προτάσεις για να βελτιώνονται οι καταστάσεις και να ευνοούνται οι συγκλήσεις. Το είπε και ο συνάδελφό μα από τη Δανία Ευρωβουλευτή, ότι ορισμένοι δείκτε είναι ανεπαρκεί. Επίση, σημειώνω ότι πολλοί συνάδελφοι καλωσορίζουν αυτή τη διαδικασία βεβαίως ε, θέλοντα πάντα να διατηρήσουν τι εξουσίες και τι αρμοδιότητε και τα προνόμια των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι θεμητό αυτό, και προτείνουν να εμβαθύνουμε τη συζήτηση και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, το είπε ο συνάδελφο από την Πορτογαλία. Για να ανοίξουμε όμω ταυτόχρονα τη συζήτηση για τον τρόπο και την επιλογή των μέσων. Ο συνάδελφος από την Αυστρία επέμεινε ότι ε, αυτό θα πρέπει να είναι σε εθνικό επίπεδο. Ναι, δεν είναι λάθος αυτό, αλλά δεν μπορούμε ε, να αφαιρέσουμε κάθε ουσία από την ε, άσκηση αυτής συντονισμού για προτάσεις. Βεβαίως η πρωτοβουλία των μέτρων που θα ακολουθηθούν και των οδών παραμένει στα κράτη-μέλη, αλλά κάποιες προτάσεις μπορούν να γίνονται. Γενικά εκφράσατε την επιθυμία και συμφωνούμε και εμείς στο Κοινοβούλιο να ε, μπούμε σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, να είναι πιο συγκεκριμένες οι συστάσεις και όχι η απλή επανάληψη των συνήθων θεμάτων. Να ενδιαφερόμαστε για τα ουσιαστικά ζητήματα και απέναντι σε αυτά, σε τακτές ε, περιόδους, να γίνονται αξιολογήσεις και των στόχων που έχουν τεθεί και μπορούν να αναθεωρούνται και αυτοί, ας πούμε. Ε, τα προγράμματα μεταρρυθμιστικά στην αρχή βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον προκαλούν αύξηση της ανεργίας και είναι λυπηρό αυτό. Ε, λοιπόν, κάθε φορά να ελέγχουμε κατά πόσο είναι εύστοχες αυτές οι προσπάθειες και οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι ε, οι σωστοί, να αξιολογούμε τα αποτελέσματα και να έχουμε και ένα πιο λεπτό συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τελειώνοντας, να αφαιρθώ στο αίτημα του συναδέλφου Μαρίνη να έχουμε τακτικές επαφές και συναντήσεις και εμείς το επιθυμούμε νομίζω και ε, με κάθε φορά ένα συγκεκριμένο θέμα, όχι έτσι γενική ανταλλαγή απόψεων και σήμερα ε, η συζήτηση αποσκοπούσε σε μια γενική ε, τοποθέτηση των παρόντων για το πώς βλέπουν και αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Στις επόμενες συναντήσεις νομίζω θα πρέπει να ασχοληθούμε με πιο συγκεκριμένα θέματα όπως λέγει και ο πρόεδρος Μαρίνη, να συνεχίσουμε αυτή τη κοινή μας ε, ε, προσπάθεια προβληματισμού. Και όπως είπα στην αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία ηγεμονική ε, βλέψη, γνωρίζει τα όρια των αρμοδιοτήτων του και θέλει απλώς να συνεργαστεί αγαστά με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ όλους. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Στο μέλλον σκοπεύουμε εμείς να διοργανώνουμε δύο σημαντικές συναντήσεις με τα κοινοβούλια. Την πρώτη πριν από το Εαρινό Συμβούλιο, στα πλαίσια της λεγόμενης εβδομένης εβδομάδας και στη δεύτερη φάση μετά το καλοκαίρι για την αξιολόγηση του εξαμήνου και αυτό ακριβώς κάνουμε και σήμερα, αν θέλετε, εν μέρη τουλάχιστον. Συνεπώς σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην συζήτηση και όπως είπα προσβλέπουμε στην ενίσχυση των σχέσεών μας και στην περαιτέρω εμπλοκή των κοινοβουλίων των κρατών μελών στις δραστηριότητές μας. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες 4 και 30, ως εκ τούτου έχετε 10 λεπτά διάλειμμα. Okay. Right. We're ready to Ψηφίζουμε λοιπόν. Το MIFIR και το NIFID που ξέρετε τι είναι. Πρώτα το κανονισμό και μετά την οδηγία. Μάρκος Φέρμπερ, θες το λόγο. Ξέρω ότι κάποιο άλλο συνάδελφο θέλει. Ναι, θέλει και ο κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τους τελευταίους μήνες, σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων, εργαστήκαμε σε ένα ε, κείμενο που μας διευκόλυνε και την ψηφοφορία. Ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία, θα το δούμε, θα δείξουν οι ψηφοφορίες. Κατά τα άλλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεργάστηκαν επικοδομητικά για να μπορέσουμε σήμερα να ε, κάνουμε αυτή την ψηφοφορία. Και σας ευχαριστώ. Thank you. Robert. you oh. Euh, κύριε Σκέπελ, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Μάρκο Φέρμπερ και όλους τους άλλους σκιώδης ηγητές για την πολύ επιμελή εργασία που είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε σε πέρα στο αποτέλεσμα των συζητήσεών μας σήμερα είναι ενώπιό σα, ε, υποτύπων τροπολογιών και συμβιβαστικών. Είναι γενικά ένας ικανοποιητικό ε, ε, συμβιβασμός και η ομάδα μου μετά από πολλές αφιβολίες και αφιταντεύσει για το άρθρο 24 τελικά συμφωνεί με τους γενικού συμβιβασμού που προτείνει ο εισηγητή Μάρκο Φέρμπερ. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ομάδα μου θέλει να πάει στην Ολομέλεια και επιφυλασσόμεθα ε, του δικαιώματος να καταθέσουμε ενδεχομένω τροπολογίες μόνοι μας ή μαζί και με άλλους για ορισμένα ε, στοιχεία και πτυχές του θέματος που μπορούν να χωρέσουν ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. I don't see Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο. Ζητεί το λόγο. Να ψηφίζουμε για τον κανονισμό. Πρώτα. Α, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Ε, παρακαλώ. Και εσύ, Μάρκους, πατήστε τα κουμπιά σας. Test vote. I can't see. All oh, right. Right, there's 42 cards plugged in and 41. 42 κάρτες έχει 43 αλλά ψηφίζουν 42. Πάντα ε, κάποιο έχει βάλει κάρτα αλλά δεν ψηφίζει. Ωραία, αυτή ήταν η δοκιμαστική ψηφοφορία. 36. Ωραία. Ε, η συμβιβαστική α ψήφιπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β. Είναι αμέσως μετά. Uh, Είναι σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική σε. Είναι στη σελίδα 7 στο δικό μου κείμενο. Τη βρήκατε όλοι. Εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία που προτείνουν οι πράσινοι. Συμφωνείτε να δεχθούμε την προφορική τροπολογία. Ναι. Τι ψηφίζουμε λοιπόν. Την συμβαστική μαζί με την προφορική τροπολογία. Είναι ένα νέο συμβαστικό κείμενο. Μάρκος. Όχι, κανονικά πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την τροπολογία των πρασίνων και αν δεν εγκριθεί τότε τη συμβιβαστική σε. Ευχαριστώ. Με την προφορική ε, τροπολογία του εισήγητου. Λοιπόν, έχουμε προφορική τροπολογία των πρασίνων που συμπεριλαμβάνει μετά και προφορική του εισηγητού. Όχι, όχι. Πρώτα των πρασίνων. Υπέρ, παρακαλώ, της τροπολογία των πρασίνων, τη προφορική Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε, τι έχουμε, τη συμβαστική σε... Α, έχουμε και άλλη προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ξεχωριστή, λοιπόν. Η προφορική τροπολογία του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές Επίσης απορρίπτεται. Τσεκ, ας το ελέγξουμε. Ψήφισα τέλει. Πέρασε. Τριάντα δύο υπέρ, οκτώ κατά. Επομένως, Α, κάποιος άλλαξε γνώμη από την προηγούμενη ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν η προφορική τροπολογία και πάμε στη συμβαστική σε μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική δε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I Στη σελίδα 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ομικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ. Α, είναι σε δύο τμήματα η W. Τμήμα πρώτον, λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Ε, συμβαστική X, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ύψιλον. Α, μια στιγμή εδώ έχει ένα σωρό προφορικές αυτή. Τρεις προφορικές πρώτα τροπολογίες με τη σειρά. Η προφορική της άλτε των φιλελευθερών υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η προφορική δεύτερη πάλι των φιλελευθέρων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και η τρίτη προφορική των πρασίνων υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται. Τώρα έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές Επίσης εγκρίνεται. Α, το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική Z, Z στη σελίδα 37. Προφορική τροπολογία πρώτα, υπέρ της προφορικής κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η συμβιβαστική Z όπως ήταν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 40, συμβαστική ΑΑ. Those in favor. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τώρα, ΑΒ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΑΣ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΑΕ έχει και εδώ προφορική. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική μαζί με την προφορική υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ και πάλι με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ της κατά αποχές εγκρίνεται. Και ο συμβιβασμός μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 759 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 760 υπέρ, στη σελίδα 48 κάτω. Ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική AG υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AI ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία 97 άμα τη βρω. Θα είναι στην άλλη σελίδα 56. Λοιπόν, εδώ έχουμε προφορική τροπολογία του εισηγητή. Τη ψηφίζουμε πρώτη πέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 97 μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική IQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχω χάσει το αλφάρτο τώρα. ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AZ υπέρ... Α, κάτι ξέχασα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ. Στην ΑΖ είμαστε. Υπέρ, το πρώτο τμήμα τους. Εντάξει, κατά εποχέ εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη β' συμβιβαστική. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β, β, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. VI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι γίνεται με την 193 δεν την ψηφίζουμε. BJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Είναι ένας από το ΕΛΚ υπεράριθμος. Ξέρω τον ενθουσιασμό σας για να υποστηρίξετε τον κύριο Φέρμπερ. Ε, αλλά μπορεί κάποιος να βγάλει την κάρτα του από το ΕΛΚ. Πέρασε. 45 υπέρ, κανείς ε, κατά. Okay, now let's do it <clears throat> again for the legislative resolution. Το ίδιο για το νομοθετικό ψήφισμα τώρα, το αυτό. Vote open. We need the vote open. Sorry. Secretariat's going to sleep. Come on. Α, αποκοιμήθηκε η γραμματεία. Μην έχουμε πολύ ακόμα. Ψηφίζετε, ψηφίζετε. Άλλα πέντε κουμπιά να πατηθούν. Τρεις, δύο. Δύο. Ένας. Εντάξει. Τώρα μπορώ να πω ότι τελείωσε η ψηφοφορία. 45 υπέρ υπαψηφί, χωρίς ψήφους ε, κατά και χωρίς αποχές. Πάμε μέσω τώρα στην οδηγία. Είστε έτοιμοι για την οδηγία. Συμβιβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Συμβιβαστική C αγγλικό. Στη σελίδα 8. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική διαγλικό. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. Στη σελίδα 13 έχω την, με, την προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ πρώτα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική F και εδώ έχω προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική H, προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική H, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική J. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική και η αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική L αγγλικό στον κατάλογο. Στη σελίδα 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική N με προφορική τροπολογία. Πρώτα την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα η συμβιβαστική ΕΝ, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή και αυτή. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική όμικρον ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική π. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα έχουμε και άλλη μία προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά θέλετε να υπάρξει έλεγχος καλύτερα για την προφορική τροπολογία τώρα των πρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική Q στην 37. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική R στη σελίδα 40 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική S ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική T ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική V, υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική X ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική Y εδώ έχω προφορική τροπολογία της Γκουε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AA υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AB υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AC σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. AD τώρα. Στην σελίδα 51, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή.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 AN. Έχω προφορική τροπολογία από τους σοσιαλδημοκράτες υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική τροπολογία AN. Α, όχι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κάναμε τις δύο τελευταίες ψηφοφορίες, μην παραπονιέστε. Ε, ένα λοιπόν και με τις δύο προφορικές τροπολογίες υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική AO. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. AP μετά υπέρ κατά αποχές δεκτή AQ υπέρ κατά αποχές δεκτή AR υπέρ κατά αποχές δεκτή AS υπέρ κατά αποχές δεκτή AT υπέρ κατά αποχές δεκτή AU υπέρ κατά αποχές δεκτή AV υπέρ κατά αποχές δεκτή. AW υπέρ κατά αποχές δεκτή. AX υπέρ κατά αποχές δεκτή. AY υπέρ κατά αποχές δεκτή. AZ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά BA υπέρ κατά αποχές δεκτή. BB υπέρ κατά αποχές δεκτή, BC υπέρ κατά αποχές δεκτή, BD υπέρ κατά αποχές δεκτή, BE υπέρ κατά αποχές δεκτή, BF υπέρ κατά αποχές δεκτή, BG υπέρ κατά αποχές δεκτή, BH υπέρ κατά αποχές δεκτή, BI υπέρ κατά αποχές δεκτή, BJ υπέρ κατά αποχές δεκτή, BK υπέρ κατά, όπα, λάθος λέει η πρόεδρος, επανέρχομαι σε προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. BK λοιπόν με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. BL υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτή. BM υπέρ κατά αποχές BN υπέρ κατά αποχές δεκτή, BO υπέρ κατά αποχές δεκτή, BP υπέρ κατά αποχές δεκτή, BQ υπέρ κατά αποχές δεκτή, καλύπτεται και η 2.20, η 3 έχει αποσυρθεί, οπότε ψηφίζουμε την BR, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. BS, με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής. Κατά. Αποχές. Δεκτή η προφορική. Ψηφίζουμε την BS τώρα με την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. BT υπέρ κατά αποχές δεκτή. BU υπέρ κατά αποχές δεκτή. BV υπέρ κατά αποχές δεκτή. BW υπέρ κατά αποχές δεκτή. BX υπέρ κατά αποχές δεκτή. BY υπέρ κατά αποχές δεκτή. BZ υπέρ κατά αποχές δεκτή, CA υπέρ κατά αποχές δεκτή, CB υπέρ κατά αποχές δεκτή, CC υπέρ κατά αποχές δεκτή, CD υπέρ κατά αποχές δεκτή, CE υπέρ κατά αποχές δεκτή, CF υπέρ κατά αποχές δεκτή, CG υπέρ κατά αποχές δεκτή, Τώρα έχω κατά διέρεση ψήφο εδώ τη συμβιβαστική CH πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. CI υπέρ κατά αποχές δεκτό, CJ υπέρ κατά αποχές δεκτό, CK υπέρ κατά αποχές δεκτό, CL υπέρ κατά αποχές δεκτό, CM υπέρ κατά αποχές δεκτό, CN υπέρ κατά αποχές δεκτό, CE ο υπέρ κατά αποχές δεκτό CP υπέρ κατά αποχές δεκτό CQ υπέρ κατά αποχές δεκτό CR υπέρ κατά σε δύο τμήματα μάλλον πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ δεύτερο κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό CS υπέρ κατά αποχές δεκτό. CT υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τελική ψήφο στο τροπολογημένο πλέον κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέραν της ψηφοφορίας 44 υπέρ, κανείς κατά καμία αποχή. Και τώρα η ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίζεται. Ένας ακόμα ψηφίζει, ένας ακόμα, πέρα στις ψηφοφορίες, 44 λοιπόν, υπέρ. Μάρκος, θα ήθελες το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ θερμότατα. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν έδειχνε η υπόθεση ότι θα ήμασταν τόσο συμπαγείς και στοιχημένοι στη ψηφοφορία. Πάντως χαίρομαι που η Επιτροπή μας έχει μία γραμμή με αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες για τις χρηματαγορές, προστασία του καταναλωτού, προστασία του φορολογουμένου. Είμαστε προετοιμασμένοι για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το οποίο βέβαια δεν είναι σε θέση να διαπραγματευθεί μαζί μας. Μπορεί να υιοθετήσει το σύνολο των δικών μας προτάσεων και να τελειώνει υπόθεση. Ε, τώρα, παρόλο που είναι τόσο μονοσήμαντο το αποτέλεσμα, χρειάζεται την νομιμοποίηση και από την Ολομέλεια και θα παρακαλούσα το συντομότερο ή δυνατόν τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια για να έχουμε σαφή ε, απόφαση και να πούμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Uh, I see that Robert is nodding in agreement with that. Ola, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, όλες το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα απλώς να επενέσω τον Μάρκους και τους άλλους και όδες εισηγητές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για εξ ονόματος ολόκληρης ομάδας μου γιατί είμαστε στην πλειοψηφία αυτή τη φορά. Okay. Thank you, thank you, thank you very much. Um, so I think we have, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως έχουμε συνένεση λοιπόν. Θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Θα δούμε στην Ολομέλεια πότε θα μπει το θέμα και θα το αφήσουμε στην γραμματεία. Ζητάμε αν είναι δυνατόν να μπει τον Οκτώβριο στην ημερήσια διάταξη. Έτσι ε, ώστε να το ολοκληρώσουμε. We've got another vote somewhere. Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretariat sitting next to here. Okay. Are we, are we organized? Έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Προχωράμε στο σχέδιο έκθεσης του Σαν Ποτέρχο προς μια ενωπαϊμένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων. Να δω που είναι ο εισηγητή. Αν χρειαστεί βοήθεια κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία. Είστε όλοι έτοιμοι. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κρίση περνάμε, κανένας δεν δείχνει τι θέλει, ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, Μπορούμε να πάμε ένα μπλοκ μέχρι και την 28. Unblock. Μα σας παρακαλώ, εντάξει, το ξέρω. Εδώ κάνετε ε, επαφές, αλλά μπας περιπτώσει μπορούμε να ψηφίσουμε unblock μέχρι την 28. Όχι, δεν θέλατε.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Ε, Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά, <clears throat> υπέρ κατά αποχές έχουμε την 39 ηλεκτρονικά. Everybody's voted, closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά πρέπει να ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 προς 15. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Every voted, votes closed. That is carried 20. Τέλος εγκρίνεται 22 υπέρ 21 κατά. Πού και πού τα καταφέρνω. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 59 υπέρ τι λέει Okay. 59 Ψηφίζουμε την 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, οπότε μάλλον προτιμάμε την ΙΜΚΟ 14. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58. Φαντάζομαι πως είναι συμβατή. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ Υπέρ, κα... υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 15. Υπέρ. Έχουμε την ΙΜΚΟ 15. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα το ελέγξω, αλλά νομίζω αυτό είναι ο συνδυασμός 22-21. probably wrong now. we are, 22-21. 22-21, υπέρ. 69. Όχι. Α, F. Ωραία. Συμβιβαστική F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Αυτό θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 σε πέρι, 22 κατά. Καταπίπτει. Λοιπόν, απορρίπτεται 82 υπέρ κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα, συγγνώμη, το τρίτο τμήμα είμαστε. Τρίτο τμήμα της συμβαστικής G, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 20 με 23. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Μα τι είναι αυτό. Okay. 82. All those in favor, against abstentions, that's carried. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε για την, ηλεκτρονικά για την 83. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 23 κατά. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H σε διάφορα τμήματα. 4. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 17 υπέρ, 26 κατά. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε και πάλι. τώρα είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και το τέταρτο τμήμα υπέρ κατά θα ελέγξουμε πάλι. Ε, γίνεται δεκτή. Προχωράμε στην 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ 98 96 και 97 ε, ήταν οι ίδιες. Έχετε δίκιο, πάμε στην 99. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 99. Right, votes closed. That's rejected. 21. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε. 104. Κάποιος ακόμα. Όχι. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία. Καταπίπτει. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΜΜΑ. σε δύο τμήματα. Η πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Votes closed. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 προς 21 ψήφι. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π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 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έπειτα, οι παραπομπές μέχρι και τη 14 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική τάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. votes closed. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 22 προς 21 ψήφους. Η τροπολογία 5. υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο Εκτιμώντας β, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο εκτιμώντας γ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16, γιατί 16. Α, εγώ είμαι στην 18. 16. 16. Πέρασε η 16. Λοιπόν, 17 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε για το κείμενο όπως τροποποιηθήκε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 υπέρ, κανένα κατά και 22 αποχές. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τον εισηγητή. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα, οπότε επόμενη συνεδρίαση είναι Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 3.